χαμηλής ε, ανάκαμψης, ανοίγματα νέων αγορών είναι σημαντικά. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη στήριξη σας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λοιπόν δύο προτάσεις ψηφίσματος για να κλείσουμε τη συζήτηση που θα ψηφιστούν αύριο στις 12. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε σε μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή για την αύξηση των νορβηγικών δασμών για κάποια ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μορέιρα που έχει επιβάλει την ερώτηση για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Αυτή η ερώτηση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εμπορίου, Διεθνού Εμπορίου που είμαι πρόεδρος της στην Ευρωβουλή και υπό αυτό τον όρο είμαστε εκπρόσωποι αυτής της ερώτησης πάλι και εξ ονόματος από του Ευρωβουλευτή του Κρίστοφ ε, Φιέρνερ που προσυπογράφει. Το κείμενο αφορά το ότι από τον Ιανουάριο 2013 η εξαγωγή ε, ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένων κρεάτων, βοήου κρέατος για παράδειγμα, ε, υφίστανται τέλη ε, και δασμούς ε, τελωνιακούς ε, σε σχέση με 334% αύξηση όσον αφορά την νορβηγική αγορά. Ερώτηση λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, υπήρξε διαβούλευση, ενημερώθηκε για αυτή την πρωτοβουλία, για αυτά τα προστατευτικά μέτρα της Νορβηγίας και για τις επιπτώσεις αυτών των μέτρων όσον αφορά τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Νορβηγία σε αυτά τα προϊόντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει παραβίαση ή όχι των υποχρεώσεων της Νορβηγίας όσον αφορά τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και για την συμφωνία από πλευρά της ε, ε, Νορβηγίας ε, για την χορήγηση ειδικών δυνατοτήτων για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι πρόκειται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το να υπάρξουν αξιόπιστες πρόοδοι όσον αφορά την κυβέρνηση της Νορβηγίας για να επιληθεί το ζήτημα αυτό. Αυτό είναι το κείμενο της ερώτησης. Και γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτούς τους λόγους ενδιαφερόμαστε άμεσα να γνωρίσουμε ποιες είναι οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτές τις ερωτήσεις. Επιτρέψτε μου δύο σκέψεις από πλευράς μου. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούται να ακολουθεί μια πολιτική ε, εμπορικού ανοίγματο. Πάντα καταγγέλαμε τα, μέτρα, τα προστατευτικά μέτρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ιδιαίτερα ισχύει αυτό με χώρε που έχουμε συμφωνίε εταιρική σχέση, όπω με την Νορβηγία, μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ιδιαίτερα. Δεύτερον, και σε σχέση με το, τα επιχειρήματα αυτά. Οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγίας είναι ιδιαίτερα ισχυροί, ισχυρές. Είναι ο πρώτος εταίρος εμπορικά της Νορβηγίας η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε και προσπάθειες που καταβάλλονται για μια σταδιακή απελευθέρωση μέσα στο πλαίσιο των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων. Τώρα λαμβάνονται νέα προστατευτικά μέτρα από πλευρά της Νορβηγίας σε σχέση με το εμπόριο μεταξύ των χωρών μας και αυτό είναι μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους και πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της απελευθέρωσης ε, του τομέα αυτού ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένουμε τις απαντήσεις κατεπηγόντως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Επίτροπος έχει τον λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξη που παρέχει ε, σε σχέση με τα μέτρα που πήραμε για την Νορβηγία. Είναι ε, καλοδεχούμενα τα σχολεία σας. Ε, τα μέτρα τα οποία έλαβε η Νορβηγία είναι προστατευτικού χαρακτήρα. Δεν είναι το είδος της δράσης που θα ανέμενε κανείς από την φίλη και γειτονική αυτή χώρα. Λυπούμε που αναφέρω ότι δεν είχε διαβουλεύσεις μαζί μας, δεν συνοήθηκε μαζί μας η Νορβηγική κυβέρνηση πριν προχωρήσει στην αύξηση των δασμών. Αφού η απόφαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε όλα τα απαραίτητα και διαθέσιμα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτή τη ε, κρίση. Ο Γενικό Διευθυντή τη ΓΔΑ, ο Επίτροπο ε, Τσιόλο, εκφράστηκαν κατά των νέων δασμών. Έγιναν διαβουλεύσει ε, σε πολιτικό τεχνικό επίπεδο με την Νορβηγία. Ετέθη το θέμα και στην Κοινή Επιτροπή αλλά δεν μπόρεσε, δεν έλαβε υπόψη της η Νορβηγία ούτε και επανεξέτασε ή αναθεώρησε αυτά τα μέτρα. Θα πρέπει να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτών των δασμών και τελών που μάλλον θα είναι ε, μέτριος για τους πρώτους μήνες 2013. Οι εξαγωγές τυριού ε, αυξήθηκαν κατά 1,5% ε, προς την Νορβηγία παρά τους αυξημένους δασμούς. Βέβαια, μακροπρόθεσμα αυτοί οι νέοι δασμοί θα μπορούσαν να περιορίσουν την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς Νορβηγία για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι σε ό,τι αφορά τις ορτανσίες, ε, η εξαγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 3 εκατομμύρια ευρώ το 2012 έπεσαν στο 1 εκατομμύριο ευρώ το 2013 μετά ε, την αλλαγή ταξινόμησης στο πλαίσιο του τελωνιακού ε, κώδικα. Έχουμε το άρθρο 19 της Συμφωνίας για την Οικονομική Εταιρική Σχέση. Έχουμε και τις διμερείς συμφωνίες και τα άρθρο 19 αυτής της συμφωνίας, τα οποία προβλέπουν προοδευτική εμπερική, εμπερική απελευθέρωση τα άρθρα αυτά. Και είναι και στι δεσμεύσει τη Νορβηγία στο πλαίσιο του ΠΟΕΦΑ. πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε διμερό. Θα λάβουμε υπόψη ε, βέβαια το θέμα αυτό και σε άλλου τομεί ε, τη σχέση μα με την Νορβηγία. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ, Επίτροπε. Για δύο λεπτά θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Στάσνη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η θέσπιση δασμών για την εισαγωγή οργικών προϊόντων αποτελεί κατάφορη παραβίαση ε, των διμερών συμφωνών και όσον αφορά το γράμμα και όσον αφορά το πνεύμα. Τα μέτρα αυτά της Νορβηγίας πρέπει να θεωρηθούν προστατευτικά και απαγορευτικά προς το εμπόριο. Είναι μια απόφαση η οποία αντιβαίνει σε μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την αρχή της απελευθέρωσης του εμπορίου. Η Νορβηγία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης θα πρέπει να σέβεται, δεσμεύεται στο ότι θα σέβεται αυτές τις αρχές. Από την άλλη πλευρά αυτοί οι περιορισμοί εγκρίθηκαν χωρίς να προηγηθεί καμία διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι απαράδεκτο διότι η Νορβηγία είναι μια χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στενότατος οικονομικούς ε, και πολιτικούς δεσμούς. Είναι επίσης ακατανόητο το πώς μια χώρα που απέφυγε τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης θέλει να θεσπίσει τέτοια μέτρα. Εμείς στην Επιτροπή ΙΝΤΑ καλούμε την Νορβηγική Κυβέρνηση να αποσύρει τα μέτρα και να ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα για την επίλυση του ζητήματος. Προσωπικά ελπίζω, ελπίζω ειλικρινά ότι αυτές, ε, αυτοί οι αστρονομικοί δασμοί που ξεπερνάνε το 200, 300, το 400% θα είναι κάτι που δεν το ξαναδούμε ποτέ σε αυτή την ε, περιοχή. Ιδίω με έναν τόσο στενό εμπορικό εταίρο για μας όπως είναι η Νορβηγία. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σερτούγκα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Παγκόσμια, ιδιαίτερα στον χώρο του γύρου της Ντόχα, ζητούν να υπάρχει λιγότερο, μικρότερο προστατευτικό πλαίσιο για τις, τα γεωργικά προϊόντα στις αγροτικές αγορές. Έχουμε όμως χώρες με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και εν μέρη με μεγάλη εξάρτηση από τη γεωργία και με μεγάλη επιφύλαξη πρέπει να αντιμετωπιστούν τα θέματα της απελευθέρωσης. Μόνο που η Νορβηγία είναι μια πολύ ανεπτυγμένη χώρα στην Ευρώπη με συγκριτικά μικρό γεωργικό τομέα και σε σχέση με τα όσα έγιναν στο 2011 με την κρίση του βούτυρου με υψηλότατες τιμές ε, έχουν ε, αφήσει τα ίχνη και σε σχέση και με το λαθρεμπόριο που αναπτύχθηκε και ε, επιβαρύνθηκε ο πληθυσμός της Νορβηγίας. Τώρα για τις μικρές επιχειρήσεις, μικρές εκμεταλλεύσεις που δεν είναι ίσως ανταγωνιστικές και που δεν θέλουν να εκτεθούν στην ανταγωνιστική πίεση της απελευθερωμένη αγοράς, όμως θα πρέπει να βρει άλλο τρόπο η Νορβηγία από τους υψηλότατους αυτούς δασμούς που επιβάλλει στα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω δύο ερωτήσεις, Επίτροπε. Τη μία την απαντήσατε. Θα ήθελα να ξέρω τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τούδε. Αυτό το επεξηγήσατε σύντομα. Αλλά επίσης ε, και σε σχέση με διμερείς επαφές, ε, πώς κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει όπως αναφέρθηκε σε διμερείς επαφές και σε σχέση με τους νορβηγούς ε, εταίρους, πώς μπορείτε να τους πείσετε να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα για να προστατεύσουν τους γεωργούς τους αντί τους υψηλότατους αυτούς δασμούς. Ευχαριστώ. Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε. Ήμουν εισηγητής στην γνωμοδότηση για την Γεωργική Επιτροπή για την ε, εμπορία με γεωργικών προϊόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας και στη διμερή εμπορική συμφωνία εντάχθηκε η γνωμοδότησή μας το 2012. Στη συμφωνία αυτή και τα δύο μέρη είχαν αναλάβει την υποχρέωση να συνεχίσουν με το πνεύμα του άρθρου 19 της συμφωνίας ΕΟΧ. Και στη συμφωνία αυτή τα δύο μέρη δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες έτσι ώστε να έχουμε προοδευτική απελευθέρωση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων. Και μετά έλεγε πως το 2014 θα γινόταν μια αναθεώρηση των εμπορικών συνθήκων έτσι ώστε να διερευνηθούν κάποιες ενδεχόμενες ε, περαιτέρω παραχωρήσεις. Αυτή ήταν μια συμφωνία την οποία είχαν υπογράψει και οι δύο πλευρές τότε γιατί ήταν σε εισαγωγικά αμοιβαία συμφέρουσα. Αυτή τη στιγμή η η εμπορική αυτή, η εμπορία γεωργικών ε, προϊόντων με την Νορβηγία είναι το 5,9% των εξαγωγών τους και το 10% των εισαγωγών τους. Και μου κάνει εντύπωση λοιπόν που ακολουθούν αυτή την τακτική που αντιβαίνει με τα όσα συμφωνήθηκαν. Εγώ θα ήθελα να παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει δράση για να μειωθούν αυτοί οι δασμοί πριν την επόμενη αναθεώρηση που θα γίνει το 2014. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Άσουαρ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Μπέντσεν. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πριν από κάποιες εβδομάδες η νορβηγική κυβέρνηση αύξησε τους δασμούς από μηδενικό επίπεδο σε πάνω από 250%. Αυξήθηκαν λοιπόν σε δυσθεώρητα ύψη. Το ίδιο ισχύει και για τα τυριά και για το πρόβιο κρέας για το πρόβιο πάνω από 300%. Λοιπόν, η Νορβηγία δεν είναι μια φτωχή χώρα, είναι μια πλούσια χώρα που έχει τεράστιο ε, πλεόνασμα στο εμπορικό της ισοζύγιο. Και παράλληλα με αυτό υπάρχει και η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό, Χώρο που με το αντίστοιχο άρθρο γίνεται λόγος για απελευθέρωση του εμπορικού πλαισίου. Από το 2012 αυτό άρχισε να ισχύει, δηλαδή πρόσφατα σχετικά. Και οι δύο αμφότερες πλευρές, το τονίζω αυτό, αμφότερες οι πλευρές θα λαμβάνουν μέτρα ώστε να μεριμνούν και να διασφαλίζουν ότι τα προτερήματα θα είναι αμοιβαία από αυτή την δράση τους ε, και δεν θα διαμφισβητούνται ή δεν θα υπονομεύονται. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό που συμβαίνει τώρα από τους Νορβηγούς είναι ακριβώς το αντίθετο αυτού που διασφαλίζει αυτό το άρθρο. Τώρα μπορώ να κατανοήσω βέβαια πρέπει να πω ότι το εμπόριο με ε, γεωργικά προϊόντα μπορεί να μην διαδραματίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο το εμπόριο με τα ε, ψάρια ή άλλα σημαντικά θέματα για την Νορβηγία. Κατανοώ ότι θέλει να διασφαλίσει το βιωτικό της επίπεδο η Νορβηγία, αλλά δεν κατανοούμε καθόλου τη, αυτά τα μέτρα και τη σκοπιμότητά τους. Ελπίζουμε ότι αύριο θα αποσταλεί ένα σαφέστατο μήνυμα προς την νορβηγική κυβέρνηση ότι είμαστε κατά, κάθετα, κατά του προστατευτισμού και ότι δεν είμαστε σύμφωνοι με κανένα τρόπο στο ότι δεν υπήρξαν διαβουλεύσεις προτού ληφθούν αυτά τα μέτρα. Είναι απαράδεκτα αυτά τα μέτρα και αυτή η κατάσταση στην οποία κατέληξε η Νορβηγία. Και γι' αυτό απευθύνω έκκληση και ζητώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει πραγματικά σθένος σε αυτό το θέμα. Να πιέσει και να απαιτήσει να, και να μας πει τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναντι αυτού του προστατευτικού μέτρου που έλαβε η Νορβηγία. Τελάνγκια για να τελειώσουμε για δύο Πρέπει να σας πω κύριε Πίτροπε πως έχουμε μια ωραία παροιμία στα Ολλανδικά που λέει δεν θα πρέπει κανείς να ροκανίζει το τυρί που έχει στη φρυγανιά. Τι σημαίνει αυτό. Πώς θα πρέπει να στηρίζουμε τις θέσεις που έχουμε υπογράψει και να μην αφήσουμε την Νορβηγία να μας φάει το τυρί από το ψωμί που έχουμε μπροστά μας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 Καταλαβαίνετε πως αυτοί οι τεράστιοι δασμοί που επιβλήθηκαν δεν μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της αμοιβαίας συμφωνίας από τη μία μέρα στην άλλη. Για τις ορτανσίες που φεύγουν από την Ολλανδία για παράδειγμα ε, ήταν κάτι το αδιανόητο. Το γκούντα το τυρί δυόμιση φορές επάνω. Μπορεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως αυτό δεν είναι ε, φοβερό γιατί δεν είναι ο βασικός μας εμπορικός εταίρος αλλά στη δική μου εκλογική περιφέρεια πέρα να σας πω ότι έκλεισαν επιχειρήσει από αυτό. Τόσο απλό είναι. Αν η Νορβηγία θέλει να έχει πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές, θα πρέπει και εμείς να έχουμε πρόσβαση στις νορβηγικές αγορές και ξέρετε πως αυτά τα εμπόδια τα εμπορικά ισχύουν εδώ και μήνες και προκαταρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν έχει κάνει κάτι το πολύ συγκεκριμένο. Νομίζω πως θα πρέπει να επιμείνουμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει την Ορβηγία έτσι ώστε πολύ σύντομα να ξεκινήσουν σε υψηλό επίπεδο διαπραγματεύσεις για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπορικά εμπόδια και αν δεν συνεργαστούν οι Νορβηγοί να λάβουμε μέτρα κατασταλτικά για παράδειγμα, ενδεχομένως εναντίον του νορβηγικού σολομού. Έτσι ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να έχουμε μία ισόρροπη σχέση με την φίλη χώρα Νορβηγία. Αλλά εντωμεταξύ ας μην τους αφήσουμε να μας αρπάξουν το φαΐ από το πιάτο. Ε, ελπίζω ότι αυτό θα σημεί με τη βοήθεια της Κομισιόν. Θα δώσω τώρα στον Επίτροπο το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους ε, βουλευτές του Κοινοβουλίου που έθεσαν το ζήτημα αυτό. Να σας ευχαριστήσω για τα αποφασιστικά σας λόγια, για την όλη συζήτηση. Ε, λαμβάνω υπόψη μου τα όσα είπε ο κύριος Ερτούκ, αλλά και άλλοι για την αναθεώρηση των ε, εμπορικών όρων. Αυτό προβλέπεται, το πώς είπε και ένας άλλος συνάδελφος, για το 2013-2014 και αυτό θα πρέπει να οδηγήσει στο άνοιγμα ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων με στόχο την περαιτέρω απελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την πολιτική υποστήριξη που θα μας παράσχεται αν αύριο με μεγάλη πλειοψηφία το ψήφισμα. Θα σας διαβεβαιώσω ότι θα το λάβουμε υπόψη, όπως ε, ε, είπα και πριν, σε άλλους τομείς και σε άλλες πτυχές των σχέσεων μας με την Νορβηγία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος ε, που θα κλείσει τη συζήτηση, η οποία ολοκληρώνεται τώρα και αύριο θα λάβει χώρα η ψηφοφορία στις 24 ε, Ιουλίου συνεχίζεται η συνεδρίασή μας, έχει δημοσιευθεί η μερίσια διάταξη και στην ιστοσελίδα